Right, good morning. Καλή σα μέρα κύριε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. καλώ ήρθατε στη σημερινή συνεδρίαση τη Επιτροπή Εξωτερικών, θέμα υπαριθμών ένα τη σημερινή διάταξη που προβλέπει την έγκρισή τη. Σχόλια, όχι. Καλώ εγκρίνεται. Θέμα 2. Ανακοινώσει δεν έχω και άρα Πάμε στο υπαριθμό 3 έγκριση των πρακτικών της ε, προηγούμενης συνεδριάσεως της 11ης Σεπτεμβρίου έχουμε ήδη. Εάν δεν έχετε σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως θα θεωρήσω ότι εγκρίνεται και τα πρακτικά. Και τώρα το 4 για άλλη μια φορά καλωσορίζουμε τον πρέσβη Βάλεντε Αλμέιδα ο οποίος είναι πάντοτε προσκεκτημένος ε, στην Επιτροπή μας, εκπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη. Ως γνωρίζετε κύριε Πρέσβη, το έργο της Επιτροπής Εξωτερικών σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη βασίζεται σε ένα τρίπτυχο συστάσεις προς το Συμβούλιο για τη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με φετινό εισηγητή τον κύριο Φρόιντ που επίσης είναι εδώ δεύτερο επίσκεψη στο ε, Αρχηγείο των Ηνωμένων Εθνών και τέλος ομάδα εργασίας που εργάζεται για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών με επικεφαλή στην κυρία Μπάρβαρα Ροχ Μπίλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για την στήριξη που προσφέρατε στην ε, επίσκεψή μας τον περασμένο Οκτώβριο και η οποία πετέλεσε πραγματική επιτυχία. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή συζήτηση όχι μόνο εγώ αλλά όλοι <clears throat> θα ακούσουμε ευχαρίστως την ε, έκθεσή σας για την πρόοδο των ε, μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ κ. Γκουτιέρες και ιδίως ό,τι αφορά το πλαίσιο των περικοπών προϋπολογισμού που έχουν ανακοινώσει οι ΗΠΑ ήδη από τα τέλη του 2017. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για την κατάσταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και για το Brexit. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε είναι μεγάλη ευχαρίστησή μου να είμαι εδώ μαζί σας. Είναι και καθήκον μου βεβαίως να έρχομαι στις Βρυξέλλες και να σας συναντώ σε αυτή την πολύ σημαντική 8η Μαρτίου. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ ιδίως τις γυναίκες ευρωβουλευτές και βεβαίως και τις υπαλλήλους της Γραμματείας και όλες τις άλλες κυρίες που βρίσκονται στην αίθουσα για την σημερινή μέρα τους στη Νέα Υόρκη εργαζόμεθα ενεργά υπέρ θεμάτων ισότητας των φύλων και έχουμε και έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών την επόμενη εβδομάδα. Και η ομάδα μου εμπλέκεται ενεργά στην σύνταξη του κειμένου. Και με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχθηκα την αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας πέρσι, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, γιατί για μας είναι και το αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του έτους, διότι μας ενημερώνετε και εσείς για την κατάσταση στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το πολιτικό κλίμα όπως διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Και εμείς βοηθούμε να κατανοήσετε το τι συμβαίνει στην Νέα Υόρκη. Βεβαίω και με τον κύριο Φρόιντ για την εργασία του, καθώς και με την κυρία Λόχ Μπίλερ, την οποία θα δούμε σε λίγες εβδομάδες, ως εισαγωγική παρατήρηση στο θέμα μας, να σας πω ότι στη Νέα Υόρκη είναι πολύ ενδιαφέροντες οι καιροί που περνούμε τώρα. Διαμορφώνεται μια παγκόσμια κατάσταση ασφαλώς όχι εύκολη, ασταθής, δύσκολα διαχειρίσιμη, αλλά στα Ηνωμένα Έθνη έχουμε και καινούργιο γενικό γραμματέα. Ευρωπαίο, Πορτογάλο, επίσης, και ένας δυναμικός άνθρωπος με τα βλέμματα στραμμένα στο μέλλον. Αυτά στην Νέα παρόλα τα προβλήματα, παρόλη την ασταθή παγκόσμια κατάσταση. Βλέπω ωστόσο μια νέα ορμή μέσα στα Ηνωμένα Έθνη και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που αυτή τη νέα ορμή, τη νέα πνοή δίνει ιδίω ένα Ευρωπαίο Γενικό Γραμματέα. Πώ θα χαρακτηρίζει την κατάσταση σήμερα, Νέα ορμή, αλλά και νέε απειλέ κατά τη ε, πολυμερού συνεργασίας. και χρειαζόμαστε συμμαχίε, αλλά απειλέ έρχονται και από αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και από άλλους. Ο συνδυασμό των δύο αυτών παραγόντων κάνει την κατάσταση, όπως είπα, δύσκολα διαχειρίσιμη. Βλέπω και νέα, χάσματα να επανέρχονται. Βλέπω ένα Συμβούλιο Ασφαλείας σχεδόν σε παράδειση ανίκανο να φτάσει σε συνενέσεις για κέρια θέματα, για σοβαρές απειλές σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπω την συμπεριφορά των Αμερικανών φίλων μας τους τελευταίους μήνες και που καμιά φορά η στάση τους αυτή καθιστά τη συνένεση μεταξύ ημών και αυτών πολύ δύσκολη. Βλέπω άλλο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας την Ρωσία να προχωρεί σε τακτικές περισσότερο προσεγγίσεις αντί για πιο μακροπρόθεσμες ε, στρατηγικές προσεγγίσεις και βλέπω και την Κίνα να απλώνεται και μέσα σε αυτά τα πλαίσια βλέπω να ανοίγεται κάποιο περιθώριο και κάποιες ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση νέες ευθύνε. όπου κάποιοι αποχωρούν πολλοί θα ήθελαν να δουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εισέρχεται. Ε, έχουμε την ικανότητα να το πράξουμε αυτό, έχουμε και την διάθεση. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση σήμερα. Ο απολογισμός που κάνω μετά από λίγο περισσότερα από δύο χρόνια στην θέση μου, μετά από πολλά χρόνια βέβαια στην ε, Ουάσιγκτον ω πρέσβη στις ΗΠΑ. Ο απολογισμό μου είναι ότι στη Νέα Υόρκη, σε αυτό το πολυεθνές πεδίο, πρέπει να βελτιώσουμε το καθεστώς μας, τη δυνατότητα να δρούμε, να αντιδρούμε την αξιοπιστία μας και την επιρροή μας μέσα σε αυτό το πολυμερές ε, σύστημα. Και βεβαίω αυτό έχει επιτευχθεί, αλλά όχι χάρη σε μένα. Δεν λέω αυτό, αλλά πρώτα χάρη στην συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεύτερο, διότι αυτό οφείλεται στην δράση τη ΥΠΑ της εκπροσώπου κ. Μογκερίνη. Και επίση, διότι και σε άλλα θεσμικά όργανα και σε τούτο εδώ το Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη δική σα Επιτροπή, έχουμε ανθρώπου με μακροπρόθεσμα οράματα που κατανοούν ένα απλό γεγονό. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμο, το σύστημα πολυμερίου συνεργασία, εάν δεν είμαστε ενωμένοι. Η ενότητα είναι η αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκεί επιρροή και να καταλάβει τον χώρο από τον οποίο αποχωρούν άλλοι και που θα πρέπει εμείς να καταλάβουμε αν θέλουμε όντως να προωθήσουμε και τις αξίες και τα συμφέροντά μας. Το 2017 ήταν καλύτερο από το 2016 και είμαστε περισσότερο ενωμένοι συνολικά. Αυτό Σημαίνει πολλή δουλειά και στην Νέα αλλά πολλή δουλειά και εδώ. Και με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, το τοπίο εμφανίζεται πολύ ικανοποιητικό. Το πρόβλημα είναι οι βέβαια. Όταν είμαστε προφανώς διαιρεμένοι, αυτό έχει βαρύτατες συνέπειες στην αξιοπιστία μας. Πάτε την κατάσταση σχετικά με το ψήφισμα για την Ιερουσαλήμ. Αυτό έκανε μεγάλη ζημιά, ότι δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε δηλαδή την ενότητα στην αντίθεσή μας σε ένα ζήτημα το οποίο ευθυγραμμίζεται απολύτω με κοινέ θέσει που έχουμε και βεβαίω και με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία. Βλέπω στοιχεία διαίρεση και για το μεταναστευτικό. Και τώρα που μιλούμε, ενώ εμπλεκόμεθα σε μια πολύ σημαντική συζήτηση για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε διαιρεμένοι. Αν θέλουμε να έχει κάποια επίπτωση η συμμετοχή μας σε αυτό το Global Compact το οποίο έχουμε ζητήσει, διότι πιστεύουμε ότι η μετανάστευση δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μια ευρωπαϊκή μόνο πραγματικότητα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο θα το έχουμε για πολύ καιρό και το οποίο απαιτεί παγκόσμιες λύσεις. Αν θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε αυτές τις παγκόσμιες λύσεις, μπορούμε να έχουμε τέτοια επιρροή αν είμαστε ενωμένοι. Αν δεν είμαστε, ε, τότε θα υπαγορεύουν άλλοι το τι θα γίνει. Τώρα, Συρία και μεταρρυθμίσεις, πριν ακούσω τις ερωτήσεις σας. Για τη Συρία, δύο πράγματα, δύο επίπεδα αναλύσεως. Το πρώτο το πολιτικό επίπεδο, το δεύτερο το ανθρωπιστικό και το τρίτο το χημικό. Σε καμιά από αυτές τις πίστες ας πούμε τα πράγματα δεν είναι καλά. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω καλύτερα νέα αλλά δεν μπορώ. Στο πολιτικό επίπεδο μπλοκάρισμα, αδιέξοδο. Δεν λειτουργεί. Τα όσα έχουμε επιτύχει ως τώρα είναι να κρατήσουμε το θέμα μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα στην διαδικασία της Γενέβης της οποίας ηγούνται τα Ηνωμένα Έθνη. Μπορέσαμε να το κρατήσουμε εκεί και χάρη στην πάρα πολύ σημαντική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και με την σαφή στήριξη του Γενικού Γραμματέως. Όμως δεν έχουμε ακόμα επιτύχει να φτιάξουμε τις συνθήκες για μια πολιτική λύση στη Συρία. Και κυρίως διότι αρνούνται οι Συριακές αρχές να συμμετάσχουν σε μια σοβαρή προσπάθεια εξέβρεσης πολιτικής λύσης. Αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν τη Δαμασκό αντικειμενικά δεν πράττουν αρκετά για να την πείσουν να συμμετάσχει. στο ανθρωπιστικό επίπεδο η κατάσταση είναι σχεδόν καταστροφική. Χθες διαβουλεύθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας για τα θέματα αυτά ενέκριναν ψήφισμα προ εβδομάδων το οποίο θεσπίζει ανακοχή η οποία όμως δεν γίνεται σεβαστή για να δώσουν δίωδο για ανθρωπιστική βοήθεια αυτή μετέφθη με πολύ μερικό τρόπο και αυτό που αντελήφθησαν εχθέ είναι ότι το ψήφισμα στην ουσία δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του ο ένας ρίχνει το βάρος στον άλλο. Να μην σας πω τις ε, πιο άσχημες λεπτομέρειες από αυτό το blame game. Πιο συγκεκριμένα, οι τελευταίες πληροφορίες που διαθέτω λένε ότι η εφοδιοπομπή που θα είχε πρόσβαση ε, στην περιοχή που αποτελούσε το αντικείμενο της προσπάθειας αυτής και η οποία αποτελείται από 26 φορτηγά αυτοκίνητα, 10 από αυτά δεν ξεφορτώθηκαν καθόλου. Τέσσερα μόνο εν μέρη. Ούτε μία ιατρικού χαρακτήρα εκένωση δεν έγινε. Και τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι αναμένουν να εκενωθούν για ιατρικούς λόγους. Άρα στο ανθρωπιστικό επίπεδο δεν, δεν γίνονται και σπουδαία πράγματα. Και ξαναλέω, το ψήφισμα δεν εφαρμόζεται. Για τα χημικά που είναι σημαντικό ζήτημα στην Συριακή κρίση πάλι αδιέξοδο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν βλέπουμε πρόοδο, τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον, για τη δημιουργία συνθήκων για πλήρη λογοδοσία για την χρήση χημικών όπλων στην Συριακή σύγκρουση. Για τις μεταρρυθμίσεις ο Γενικός Γραμματεύς έχει ξεκινήσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων πάνω σε τρεις πίστες και αυτό και αυτά που προτείνει ο Αντώνιο Κουτιέρες, εάν εφαρμοστούν όλα, θα έχουμε πια ένα πολύ διαφορετικό οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εμείς υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές και ενεργά και απολύτως. Δέχθηκα σε πρόγευμα όλους τους πρέσβεις των χωρών μελών της Ένωσης την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τον Αντώνιο Κουτέρες και του εκφράσαμε την πλήρη υποστήριξή μας. Είναι δύσκολο όμω. Υπάρχει αντίσταση και εντός των ομαδεθών και εκτός για οποιασδήποτε μεταρρυθμίσει. Έως τώρα έχει γίνει κάποια πρόοδο. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε σωστή πορεία. Πλησιάζουμε ωστόσο στην καρδιά των διαπραγματεύσεων γύρω στην άνοιξη. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της υπόθεσης αυτής. Για την ώρα τα Ηνωμένα Έθνη νιώθουν την πίεση των ΗΠΑ για την μείωση των δαπανών, πιστεύουμε ότι είναι λογική, είναι και καλοδεχούμενη σε κάποιο βαθμό η πίεση αυτή. Χρειάζεται, πράγματι, χρειάζονται τα Ηνωμένα Έθνη να μπορέσουν να κάνουν τα ίδια πράγματα με λιγότερα χρήματα. Αλλά βέβαια, ξαναλέω, πρέπει να είναι λογική η πίεση των ΗΠΑ. Έω τώρα υπήρξε λογική. Δεν είδαμε υπερβολικά αρνητικέ συνέπειε τη πίεση αυτή. Το μέρο των δαπανών του προπολογισμού του ΟΗΕ έχει περικοπεί κατά περίπου 5% χωρίς να επηρεάσει την ικανότητα δράσης των ΗΠΑ. Υπάρχουν όμω σημάδια ότι οι ΗΠΑ θα ζητήσουν κι άλλα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε παίξει σημαντικό ρόλο γιατί λειτουργούμε ως γέφυρα ανάμεσα στους Αμερικανούς στην περίπτωση αυτή που θέλουν σημαντικές περικοπές και αυτούς, τους άλλους δηλαδή, που θέλουν σημαντικές αυξήσεις. Μέχρι τώρα σε όλες τις συζητήσεις περί προϋπολογισμού ε, το τελικό ε, νούμερο που δέχονται είναι αυτό που έχουμε καταθέσει εμείς στο τραπέζι. Είμαστε δηλαδή deal makers. Είμαστε αυτοί που διευκολύνουμε την τελική συμφωνία. Όλες οι χώρες μέλη έχουν αναθέσει σε μένα και στην ομάδα μου την ευθύνη των σχετικών διαπραγματεύσεων. Το θεωρώ σημάδι εμπιστοσύνης. Και βέβαια ξαναλέω, μόνο όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε τις μάχες αυτές μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Ελπίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις που ξεκινά ο Γενικό Γραμματέα, θα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να εγκριθούν, ας πω καλύτερα, από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο. Και πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία αυτή, την όρμη αυτή. Ή οδήποτε μήνυμα μου δώσετε εσείς ως ΑΦΕΤ ή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον επίγοντα χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων θα είναι καλό δεχόμενο. Αλλά και ένα μήνυμα ότι δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι επιτυχής η προσπάθεια αυτή και να μην λησμονούμε ότι συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της είναι ο μεγαλύτερος συνεισφορέας στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Ορισμένοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Όλοι μαζί είμαστε η μεγαλύτερη πηγή εισοδημάτων. Οι συνεισφορές των δικών μας χωρών μελών στον τακτικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών φτάνουν πάνω από 30% του τακτικού προπολογισμού των ΗΠΑ. Για το 2016, Τρει χώρε μέλη, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο και τα θεσμικά όργανα, ήταν μεταξύ των top 10 ατομικά, των top 10 ε, συνεισφορέων στον προπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, οι εθελοντικές συνεισφορές που είναι άλλος τρόπος χρηματοδότησης των Ηνωμένων Εθνών εκεί από τις δικές μας 28 χώρες μέλη φτάνουν περίπου το 50% του συνόλου, το, του συνόλου των συνεισφορών των 193 χωρών μελών των Ηνωμένων Εθνών. Άρα, η σχέση μας με τα Ηνωμένα Έθνη είναι, πώς το πω, απολύτως ε, συγκεραστική και σε ό,τι αφορά αξίες και αρχές αν δείτε τις δικές μας συνθήκες και τον χάρη των ΗΕ, επικαλύπτονται σχεδόν απολύτω. Και βέβαια και πάρα πολύ στενή σχέση ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή προσφέρει και τις αξίες και τα χρήματα για την πρόθεση αξιών αυτών. Θα πρέπει να είμαστε και να είστε κι εσείς υπερήφανες και υπερήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτό βέβαια σημαίνει και ευθύνες και για να μπορέσουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας μέσα σε αυτό το σύστημα πολυμερού συνεργασίας, πάλι, ξαναλέω, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Εάν το κοινοβούλιο σας μπορεί να περάσει το μήνυμα αυτό στις χώρες μέλη, πιο πολύ σε κάποιες ορισμένες από αυτές, ότι η ενότητα είναι η συνταγή της επιτυχίας, ενώ η διαίρεση σας καταδικάζει σε αδυναμία δράσης, αυτό θα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις αγωγικές παρατηρήσεις κύριε Πρέσβη. Αρκετοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε όλες τις ε, ερωτήσεις και να απαντήσετε μετά ενιαία. Ενιαία, πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι τις 10 περίπου, έχουμε λοιπόν ε, μισή ώρα και λίγο παραπάνω. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Φρόιντ, που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Σας παρακαλώ δύο-τρία λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ, Όγγεν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση κάθε φορά που σας ακούμε εδώ στις Βρυξέλλες και επίσης με μεγάλη ευχαρίστηση σας επισκεφθήκαμε και στη Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα για μένα. Γιατί επισκέφθηκα πριν από 40 χρόνια σε, με ημιεπίσημη ιδιότητα τα Ηνωμένα Έθνη. Και αυτό που ακούω έκτοτε, το μόνιμο τροπάριο, είναι μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών. 40 χρόνια τώρα το ακούω και ακόμη δεν έχω δει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά όπως είπατε, τώρα ο παρόν Γενικός Γραμματέας ε, έχει ε, τη δική του προσέγγιση για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Θα κάνω δύο ερωτήσεις και θα αφήσω τους συναδέλφους, ε, που θα είναι γενικές, θα αφήσω τους συναδέλφους να ασχοληθούν ίσως με πιο συγκεκριμένα θέματα. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μας πείτε ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφορές προσέγγισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στα Ηνωμένα Έθνη, που εσείς αντιμετωπίζετε μεταξύ, δηλαδή του συμπατριώτη σας ε, και παρόντος Γενικού Γραμματέα και του προκατόχου του, οι κύριες διαφορές, γιατί ξέρω ότι προέρχονταν από εντελώ διαφορετικά μέρη του κόσμου. Αυτό ούτως ή άλλως τους διαφοροποιεί και σε χαρακτήρα και σε προσέγγιση. Θα ήθελα ακριβώς να μου πείτε εσείς ε, πώς βλέπετε ε, να... Πώς είδατε τις μεγαλύτερες διαφορές. Και ένα δεύτερο θέμα το οποίο μόνο ακροθυγός το αναφέρατε είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ε, έχει κάπως, πώς να το πω, έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση προς τα Ηνωμένα Έθνη από τον προκάτοχό του. Και επειδή ήσασταν πρέσβης και στι Ηνωμένε Πολιτείε, την τελευταία χρονιά της Προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα θα μπορούσατε να μας πείτε με τι τρόπο έχει επηρεάσει αυτή η αλλαγή τη λειτουργία των ΗΠΑ. Η πρέσβης των ΗΠΑ, η Νίκη Χέιλι, δρά διαφορετικά, έχει άλλη προσέγγιση από τον πρόεδρο, που έχει τη δική του προσέγγιση προς τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Όγγεν, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, με, με βάση τις ομάδες τώρα, πρώτα απ' όλα η κυρία η από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Κύριε Πρέσβη. Κύριε Πρέσβη, αναφερθήκατε στο θέμα της τάσης της Κίνας στις 26 Ιανουαρίου φέτος το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ε, δημοσίευσε μία λευκή βίβλο για την ε, κινέζικη πολιτική στην Αρκτική και γενικότερα στις πολικές περιοχές. Αυτό έχει να κάνει με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη μείωση των πάγων στους πόλους. Αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση και στις βορειότερες περιοχές της Κίνας, κάτω από τον ε, Πεντηκοστό παράλληλος αυτός όμως περνάει και από την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από ό,τι άκουσα υπάρχουν κάποια σχέδια να υπάρξει και μία πολική οδός ε, του μεταξιού για να συνδεθεί η Κίνα με την Ευρώπη μέσω της βόρειας θαλασσίας οδού. Οπότε η ερώτησή μου. Αυτή η πολική ε, οδός του μεταξιού, ο πολικός δρόμος του μεταξιού συζητήθηκε καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άρνε Λίτς, ο επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ που μας έχετε ενημερώσει και για τις συναντήσεις που κάναμε στη Νέα Υόρκη οι συνεργάτες σας εκεί μας βοήθησαν πολύ. Για τη συνάντηση κορυφή του 2019 ελπίζουμε η Επιτροπή να έχει αρμοδιότητες για αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν για τους ε, στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα έχουμε αρμοδιότητα. Βεβαίως ο Γιώ Λάινεν που είναι εδώ από πλευρά Ένβη και Άφετ ασχολείται με την κλιματική ε, διπλωματία που είναι βασικό θέμα για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε πόρτες. Όπως ε, συζητήσαμε και με μια αντιπροσωπεία με το Ιράν. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ενώ έχουμε προβλήματα για άλλα θέματα με το Ιράν. Και έχουμε και τα πορίσματα των Υπουργών Εξωτερικών και έχουμε και μια έκθεση πρωτοβουλίας για τα θέματα αυτά. Θέλουμε λοιπόν να μπορέσει και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και οι μα μας να έχουν περισσότερη δράση για τα θέματα αυτά. Αλλά και το ίδιο το Κοινοβούλιο μέσω των αντιπροσωπιών του. Θα θέλαμε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε περισσότερο την δράση για την κλιματική αλλαγή και της Ένωσης και των κρατών μελών. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για την κλιματική διπλωματία μέσω της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, μέσω των πορισμάτων του Συμβουλίου, ούτως ώστε να προωθήσουμε και τους στόχους των διαφόρων ΚΟΠ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ισιά Charles Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Θαυμάσια επισκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε ως εκπρόσωπος της Ένωσης. Και συγχαίρω και την Πορτογαλία για την ε, για το διορισμό και του κύριου Κουτέρε και του κύριου Σεντενό. Αλλά μιλήσουμε τώρα για το Brexit, που είναι το θέμα που όλου μα απασχολεί, να δεν το λέμε και που θα γίνει σε ένα χρόνο. Και η Πρωθυπουργό Μέη, στην ομιλία τη στην διάσκεψη ασφαλεία και στο Μόναχο και η ανακοινώση του Συμβουλίου που διάβασα χθε, όλοι αυτοί λένε ότι θέλουν να συνεχιστεί η συνεργασία για τα θέματα εξωτερικών και ασφάλεια, ακόμη και μετά τον Brexit. Συνεργασία Ένωση Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να υπάρξει συνθήκη για την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια. Δεν ξέρω τώρα αν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν μόνο ε, διμερείς ε, συμφωνίες για ανταλλαγή στοιχείων. Τι θα γίνει όμως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή είναι η ερώτηση προς εσάς γιατί η Ένωση θα έχει μόνο μία μόνιμη θέση μετά τον Brexit. Συγκεκριμένα η Γαλλία θα εκπροσωπεί την Ένωση. Πώς βλέπετε την κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου τώρα που δεν θα είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα συντονίζεται τη στάση του με τη στάση της Γαλλίας και της Ένωσης σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν συζητήσεις γι' αυτό, για τα θέματα αυτά. Και κάτι άλλο. Είναι το θέμα της Κύπρου. Μια χώρα με την οποία εδώ και πολλά χρόνια έχω ισχυρούς δεσμούς και τη δυνατότητα να, ξανακι... να ξαναξεκινήσουν υπό τη νέα Προεδρία Αναστασιάδη οι συζητήσεις για την επανενοποίηση. Αλλά η Τουρκία βασικά πιέζει, ε, απομάκρυνε ένα ιταλικό πλοίο ε, που διερευνούσε για φυσικό αέριο. Τι δυνατότητες υπάρχουν από την αιγύδα των ΗΠΑ να ξαναξεκινήσουν αυτές τις συζητήσεις. Και για το θέμα της μεταρρύθμισης ε, των ΗΠΑ. Εγώ πάντα υποστήριζα να υπάρχουν μόνιμες θέσεις για τη Βραζιλία, την Ινδία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Υπάρχει καμία δυνατότητα να προωθεί το θέμα αυτό ιδιαίτερα από την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν σημαντικό να έχει μια μόνιμη θέση η Γερμανία χωρίς δικαίωμα βέτο. Τι δυνατότητε υπάρχουν επίση για να μην υπάρχει αυτή η κατάχρηση του βέτο από τη Ρωσία με τη στήριξη της Κίνας για την άθλια κατάσταση στη Συρία. Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για την πολυμερή προσέγγιση, είναι σαφές αυτό. Το διαπιστώσαμε τώρα που μπορεί να ξεκινήσει και εμπορικό πόλεμο και νομίζω ότι θέλει να υπονομεύσει και τον ΠΟΕ, όχι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά σε εμά που πιστεύουμε στην πολυμερή προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ, Άλντε. Ο κύριο Αουστρεβίτσιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, και εγώ να εκφράσω την ε, εκτίμηση για τη συνεργασία, την πολύ καλή που έχουμε όταν επισκεπτόμεθα τη Νέα Υόρκη, σε αποστολές προς τα Ηνωμένα Έθνη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την καλή δουλειά που κάνετε και σας παρακαλώ να συνεχίσετε και στο μέλλον. Πρόσφατα η Υποβιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επανήλθε από τη Γενέβη για την 37η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτά που ακούσαμε εκεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι θετικά. Υπάρχει μια συζήτηση στο Συμβούλιο ποια θα πρέπει να είναι προτεραιότητα ατομικά, συλλογικά, η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αντιπαράθεση με τις ε, πολιτικές για την ανάπτυξη. Πώς βλέπετε εσείς το θέμα με βάση τις συζητήσεις που γίνονται στην Νέα Υόρκη. Πώς θα περιγράφετε την κατάσταση για αυτά τα θέματα. Δεύτερον, η συνεχιζόμενη ή τουλάχιστον κάποιες συζητήσεις για την ενδεχόμενη αποστολή ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία που όπως ξέρετε πρόσφατα κατελήφθη από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ένα τμήμα της. Έχουμε ειδήσει. Τι θα προκύψει για το θέμα αυτό, τι μπορείτε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, NGL, η κυρία Σακοράφα, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την αγωνία μου για το μέλλον που προϊονίζεται για τον οργανισμό, εξαιτία, όπω είπατε και εσεί, τη συμπεριφορά ορισμένων κρατών. Καταρχήν, θα ήθελα να σα ρωτήσω την άποψή σα σχετικά με την προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Global Compass. Σα έχω ακούσει αρκετέ φορέ να υποστηρίζετε ότι τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να συνδιαμορφώσουν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση όσον αφορά το προσφυγικό ότι ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αλληλεγγύη τόσο μεταξύ των κρατών όσο και τα κράτη προ του πρόσφυγε θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των προσπαθειών αυτών. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα πρέπει να συμφωνούμε ότι από τη στιγμή που μιλάμε για ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στον πυρήνα τη θα πρέπει να τοποθετούνται κυρίω οι ευπαθεί ομάδε και μιλάω για τα συνόδευτα παιδιά που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα ήθελα επίση να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σα σχετικά με το προσχέδιο που έχει ήδη παρουσιαστεί και τι αλλάζει στην υπάρχουσα πρακτική θεωρείτε ότι με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη μέχρι σήμερα νομιμοποιείται να μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αλληλεγγύη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επειδή εσείς προηγουμένως είπατε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, πιστεύετε πραγματικά ότι μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να υπάρχουν οι προσεγγίσει, προσεγγισεις προσεγγίσεις, όταν κράτη-μέλη αρνούνται ακόμα και σήμερα να αναλάβουν έστω και το μήνυμο τη ευθύνη που του αναλογεί να, να υποδεχθούν δηλαδή αυτέ τι ευπαθεί ομάδε, όταν το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει αποφασίσει για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, γιατί ορισμένα κράτη-μέλη αρνούνται τον υποχρεωτικό διαμοιρασμό των προσφύγων, και όταν η προσφυγική σας πολιτική στηρίζεται σε μια άτυπη συμφωνία με την Τουρκία η οποία δεν στηρίζεται σε καμιά διεθνή συνθήκη που να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων. Πώς μπορούμε να συζητάμε μια χώρα υποένταξη όταν έχει βάλει παράνομα στο Αφρίν και όταν ε, αμφισβητεί διεθνείς συμφωνίες, απειλεί κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάω, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην Ελλάδα την ίδια. Εμένα όλα αυτά μου είναι λίγο αντιφατικά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. We come to our... Σας ευχαριστώ. Έχουμε στους τέσσερις τελευταίους ομιλητές. Από το ΕΛΚ πρώτα η κυρία Βοξόρ Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη που ήρθατε και για την εισήγηση που μας κάνατε. ο έλεγχος των ε, προσφυγικών ροών που διαρκώς ασκούν πίεση στα σύνορα της Ευρώπης από το 2015 ε, μας κάνουν να θυμόμαστε πως είναι αυτή μια από τις πιο σοβαρές παγκόσμιες προκλήσεις. Στην Ευρώπη έχουμε διαπιστώσει φρικτές επιθέσεις κατά των πολιτών μας και ε, ε, ως εκ τούτου θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να δεχτεί το δικαίωμα των κρατών να θέσουν σε πρώτη προτεραιότητα τα δικαιώματα των δικών τους πολιτών και επίσης να μπορούν να αποφασίζουν ποιον δέχονται στην επικράτειά τους. Η Ουγγαρία προστατεύοντας τα εξωτερικά της σύνορα έχει δεσμευθεί να προστατεύσει πλήρως και την Ευρώπη. Σωστή και συντονισμένη απάντηση στο προσφυγικό θα πρέπει να δοθεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, εδώ στην Ένωση. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε συνένεση για αυτό το θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά το κάποιο νόμιμο τρόπο μετανάστευσης ως μια επικοδομητική εναλλακτική ε, στις ε, διαρκείς αυτές ροές. Κάποιοι είναι μέρη της λύσης, κάποιοι άλλοι διαρκώς διαφωνούν. Όπως έχει δηλώσει η Ουγγρική κυβέρνηση, μια παγκόσμια συντονισμένη λύση όπως τώρα έχει ε, μάλλον συντάσσεται στη Νέα Υόρκη, δεν θα ήταν τίποτα άλλο παρά ένα κίνητρο για όλο ένα και περισσότερου ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Εμείς εδώ αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην επιτυχία της, των διαπραγματεύσεων για το Global Compact για την μετανάστευση με σεβασμό τη διεθνούς νομοθεσία και εγώ είμαι μεταξύ αυτών, Όμω ταυτόχρονα είμαι πεπισμένη ότι αν ε, ξεκινήσουμε, μάλλον να συμμετέχουμε μάλλον στις κυβερνητικές διαπραγματεύσει στον ΟΗΕ, τόσο τα κυβερνήσεις των κατορμελών όσο και η Ένωση, θα πρέπει να παραμένουμε στους εσωτερικούς μας κανόνες, ώστε να είμαστε συνεπείς. Στις 20 Φεβρουαρίου, ωστόσο, ε, ε, έγινε δήλωση σε πλήρη αντίφαση με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω κύριε Πρέσβη να εξασφαλίσετε το πλήρη σεβασμό της αρχής του κράτους δικαίου και επίσης των ευρωπαϊκών κανόνων και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται ώστε κανείς να παίρνει το λόγο σε διεθνή ε, φόρα να επιμείνετε για την εφαρμογή των συνθηκών και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών θέσεων. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. είναι ένα. Äh, Κύριε σας ε, πρέσβη, βάλτε παρακαλώ τα ακουστικά σας. Θα μιλήσω γερμανικά. Μας είπατε το 18 σε μια προηγούμενη συνάντηση θα είναι το έτος ε, των ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε πέντε μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο πρώτος Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και φυσικά και ο Γενικός Γραμματέας είναι από την Ένωση. Να δώσουμε λοιπόν το στίγμα μας. Ε, ξέρω ότι ο Τραμπ έχει επιτεθεί κατά των ενευτικών επιστολών. Ε, τι, αποστολών, συγγνώμη. Τι σημαίνει αυτό. Η ισχύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εν τη ενώση. Ο πρόεδρο Γιούγκερ ή δεν ξέρω ποιο πρότεινε ότι για θέματα εξωτερική πολιτική θα πρέπει να ψηφίζουμε κατά πλειοψηφία. Ω πρέσβη στην ε, Νέα Υόρκη το χαιρετίζετε αυτό γιατί όταν υπάρχει ψηφοφορία κατά πλειοψηφία υπάρχει και ψηφία. Τι επιπτώσει θα έχει αυτό στον ΟΕΕ. Νομίζω ότι ο συνάδελφο εδώ θα αναφερθεί στι ε, άλλε ανθρωπιστικέ ε, καταστροφέ στον κόσμο εκτό από τη Συρία. Θα αναφερθούμε και στου Ροχίνγκια όπου ήμασταν ε, πρόσφατα, αλλά θα αφήσω το συνάδελφο. Και αυτό είναι ένα δράμα. 600.000 έχουν διωχθεί από τη χώρα του. Τι κάνουν το ΕΕ. Γι' αυτό ευχαριστώ Γιολάινεν. Και να δώσω ακριβώ το λόγο στον κύριο Μπασίρ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρέζη, αναγνωρίζω τις ε, πολύ ξεκάθαρε απόψεις. Θα ήθελα να θίξω ένα-δύο πράγματα. Όπω είπε ε, και ο κύριος Αστριβίσιος πριν από λίγο, μόλι επισκεφθήκαμε τη Γενέβη και είδαμε έναν πολύ καταπονημένο ε, ειδικό απεσταλμένο εκεί τον ε, Αλχουσέιν και ένα γεγονός είναι ότι η οικονομία έχει μετακινηθεί πιο ανατολικά όπου έθνη όπως η Κίνα και η Ινδία ε, γίνονται σιγά σιγά οικονομικά πολύ ισχυρά. Αυτό είναι καλό γιατί από την απόλυτη φτώχεια μεγάλο κομμάτι του ανθρωπότητας ε, περνά σε οικονομική άνθηση. Ωστόσο, οι χώρε αυτέ έχουν ε, ε, όχι τόσο θετικά ρεκόρ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύω πω η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι απαραίτητο ότι θα οδηγήσει σε καλύτερε συνθήκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ αντιμετωπίζουμε αυτέ τι προκλήσει, πώ κερδίζουμε τον πόλεμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, δεύτερον, τα δικαιώματα των προσφύγων, τα αποτυχημένα κράτη που, όπως η Συρία, τα Αφγανιστάν, πρέπει να στηριχθούν να στηρίζονται διαρκώς ώστε να υπάρξει καλύτερη διακυβέρνηση και κράτος δικαίου και δημοκρατία και άρα να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης τα ευάλωτα κράτη όπως το Πακιστάν και η Ορδανία που ήδη είναι φτωχά καταρχάς, αυτά τα κράτη, αυτά τα έθνη τα τόσο εύθραυστα θα πρέπει επίσης να στηριχθούν ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να φιλοξενούν τα 68 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες που ζουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Να εκπαιδεύουν τα παιδιά, να προσφέρουν ε, υγειονομική περίθαλψη, εμβολιασμούς κτλ. Και να ε, διευκολύνονται έτσι τα παιδιά να περνάνε και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, πιστεύω πως θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, όντως θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Το γεγονός ότι 7 χώρες έχουν μόνο το δικαίωμα να είναι ε, είναι πολύ λιγότερο δημοκρατικό από ό,τι θα έπρεπε. Θα έπρεπε να επικρατεί πραγματική δημοκρατία. Σας ευχαριστώ κύριε Μπασίερ. Ο κύριος Σαφχάουζερ έχει ζητήσει το λόγο. Τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ίσως να μην με είδατε όταν ζήτησα το λόγο στην πρώτο γύρο. Μόνο κάποιες παρατηρήσεις έχω να κάνω. Καταρχάς, ο ΙΕ είναι ένα καταπληκτικό project το οποίο εμείς εκτιμάμε η Ευρώπη των Εθνών και των Ελευθεριών γιατί ακριβώς βρίσκεται το επίκεντρο ο διάλογος μεταξύ των κρατών. Ε, αυτό απαιτεί ε, σεβασμό μεταξύ των κρατών και σεβασμό της κυριαρχίας τους βεβαίως. Σε σχέση με αυτήν την ε, κυριαρχία ε, την έντονη παρουσία των ευρωπαϊκών κρατών θα πρέπει να έχουμε το εξή υπόψη μας. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίζεται, δεν είναι όμως απαραίτητο να έχει έδρα. Και τα κράτη πρέπει να διατηρούν την ανεξαρτησία τους. Αυτό είναι ε, σημαντικό και αναγνωρίζω ότι ο, ο πρόεδρος Τραμπ ε, βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος, στο, την ίδια οπτική έχει. Να πω και δύο λόγια για την αεροσφάλεια και την ε, άμυνα. Έχω την, θεωρώ σημαντικό ότι απέναντι στην αποτυχία του μόνου της Μινούσκα και διάφορων άλλων και δεν θα μιλήσω για τη Μινουσμά και άλλους, ε, θα πρέπει λοιπόν ε, τα μέλη της, του Συμβουλίου Ασφαλείας και πιο συγκεκριμένα η Γαλλία εκεί όπου είπα παρεμβαίνουν με κοινό τρόπο, με την αποτελεσματικότητα που έχουν να παρεμβαίνουν εκτός, ώστε να σταθεροποιούνται κάποιες ζώνες, θα ληφθούν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η θέση της ε, του εκπροσώπου της Ένωσης για να στηρίξει αυτή τη συνεργασία απέναντι στην τρομοκρατία και πιο συγκεκριμένα στην Αφρική. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και αφού έχουμε Πορτογάλο προσκεκλημένο σήμερα, τελευταία ερώτηση από Πορτογάλος. Πορτογαλίδα συνάδελφο, την Άννα Γκόμες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε πρέσβη. Το, η πιο σημαντική μεταρρύθμιση που είναι οπωσδήποτε απαραίτητη για την παγκόσμια ρύθμιση και ασφάλεια είναι η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να το προτείνει, μπορεί να το προωθεί, δεν έχω ακούσει πολλά, αλλά, αλλά εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να το βάλουμε μπρος. Και εν ώψη του Brexit θα πρέπει αυτή να είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία, ώστε να έχουμε μια μόνιμη θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όχι κάποια χώρα των, της και βεβαίως να καταργηθεί το βέτο και να υπάρχει μια, ή να περιοριστεί και να υπάρχει και μια σωστή και αναλογική αντιπροσώπευση των δυνάμεων ε, του 21ου αιώνα. Δεν ακούσατε τίποτα να λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπατε εκπρόσωπος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν ε, κάπως ε, συντονιστεί από αυτού. Δεύτερον, επειδή βεβαίως δεν έχουμε λύση για την ε, Συρία, θα πρέπει να γίνουμε λοιπόν εκεί παράγοντας και όχι απλά να πληρώνουμε. Τώρα, μετανάστευση. Λοιπόν, σα το λέω, προετοιμαστείτε για τα χειρότερα. Όπως είπε και είπατε εκπρόσωπο για τους πρόσφυγε, είπε πρέπει να αντισταθούμε στου. Ε, ε, άγριους, ε, γιατί αλλά οι άγριοι είναι και εδώ και εκτός. Το εξηβούλιο δεν κάνει τίποτα, το Κοινοβούλιο κάνει τη δουλειά του, ε, αλλά προετοιμαστείτε για τα χειρότερα. Και τέλος, η ΟΗΕ θα λάβει κάποια, κάποιο ρόλο σε αυτό το κρίσιμο σε θέμα της ε, φορολογίας γιατί εξακολουθούν να είναι ο παράδεισος των φορολογικών παραδείσων, ένας από τους παραδείσους δηλαδή, θα κάνει, θα ανακατευθείτε σε αυτό. Ξέρω ότι ενδιαφέρει και τις αφρικανικές χώρες. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεδιάντροπα ε, στάθηκε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αναπτυξιακή βοήθεια. Πού, τι, ποια είναι η θέση της ε, η ε, θέση στον ΟΗΕ. 11 παρεμβάσεις, 11 ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Έχετε 15 λεπτά να απαντήσετε σε όσο γίνεται περισσότερο. Ίσως συνάδελφοι, να σας πω για κάτι. Ότι εφόσον πάμε στη Νέα Υόρκη στα τέλη του Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ένα από τα σημεία που θα πρέπει εκεί να συζητήσουμε θα είναι οι συνέπειε του Brexit και για την δουλειά μας στον ΟΗΕ. Ήταν πολύτιμη αυτή η σύσταση. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρέσβης ε, Ντεαλμέιδα, για τις ε, ε, παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Ας αρχίσω με την πιο δύσκολη από διπλωματικό από διπλωματική άποψη η σύγκριση αυτή που μου ζητήσατε μεταξύ Κουτιέρες και Μπαν Κιμούν κανένας διπλωμάτης δεν θέλει να απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις αλλά τι θα μπορούσα να πω κάπως πιο ανεπίσημα. Σημειώνει ένα γεγονός. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι ο πρώτος πρώην Πρωθυπουργό που αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν, ε, υπήρξε Πρωθυπουργό και αρχηγός του κόμματος αρχηγός του κόμματός του ε, ε, στην πατρίδα του και βεβαίω ε, προσωπικότητα ε, διεθνή. Αυτό τον ξεχωρίζει ω προφίλ. Το άλλο είναι και δέκα χρόνια ύπατος, αρμοστή ε, αρμοστής για τους πρόσφυγες. Τα γνωρίζει τα πράγματα από μέσα και τώρα τα βλέπει και απ' έξω και αυτό του δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα Περισσότερα δεν μπορώ να πω γιατί δεν είναι αρκετά ανεπίσημο το περιβάλλον. Οι αλλαγέ τώρα των αμερικανικών θέσεων μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Έχω συνεργαστεί και με τον Πάουερ, προηγούμενο εκπρόσωπο του που είχε διορίσει ο Ομπάμα, αλλά θυμόμαι και τους παλαιότερους καιρού στα Ηνωμένα Έθνη, όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν διαφορετικέ προσεγγίσεις και στάση σε σύγκριση με αυτήν που είχε ο πρόεδρος Ομπάμα και ιδίως στη δεύτερη τετραετία του. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε τα πράγματα με κάποια απόσταση, με κάποια προοπτική. Είχαμε και άλλες περιόδους όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν πολύ, στέκονταν πολύ κριτικά απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε τώρα είναι να συνεργαστούμε όσο γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να προσπαθούμε να βρίσκουμε κοινούς τόπους συνεργασίας όσο είναι δυνατόν και υπάρχουν ακόμα πολλοί τόποι συνεργασίας. Όπου δεν μπορούμε να βρούμε όμως κοινό έδαφος, ε, τότε πρέπει να εμείνουμε εμείς στις θέσεις μας και στις αξίες μας. Και αυτό κάνουμε, κάπου τα καταφέρνουμε καλύτερα από κάπου αλλού η ανησυχία μου για την αμερικανική θέση είναι βέβαια το μήνυμα που δίνουν στον υπόλοιπο κόσμο με τον τρόπο αυτό και για κάποιους που ψάχνουν να βρουν κάλυμα έτσι ώστε να συμμετέχουν λιγότερο στα συστήματα διεθνούς συνεργασίας. Για την Κίνα και τελείως αποσυνδεδεμένο με τα όσα είπα μόλις τώρα. Για την Κίνα καθιστάμεθα μάρτυρες όπως είπα μιας διαρκώς αυξανόμενης σημασίας του ρόλου στη διεθνή συνεργασία της Κίνας και βεβαίως αυξάνει αναλογικά και με τη δημογραφία τους αλλά και με την οικονομική τους βαρύτητα. Μεγάλη λοιπόν αύξηση της σημασίας τους μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Ένας αριθμός κινέζικων πρωτοβουλειών είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Για το ιδιαίτερο σημείο που αναφέρατε για την Αρκτική δεν έχω συμμετάσχει σε οποιαδήποτε σχετική συζήτηση για την οδό του μεταξιού που περνάει από τον Πόλο αλλά ξαναλέω η πρωτοβουλία αυτή κερδίζει έδαφος μέσα στα Ηνωμένα Έθνη και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω να τοποθετηθεί σαφώς απέναντι σε αυτό το πολύ σημαντικό κινέζικο σχέδιο. Για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, εμείς ε, συμμετέχουμε πολύ και εσωτερικά και εξωτερικά και για την ανάκαμψη της αναπτυξιακής μας πολιτικής με νέα συνένεση και νομίζω ότι έχουμε και καλά χαρτιά που μπορούμε να παίξουμε. Έχουμε καλή φήμη μπορούμε ίσως να την πλασάρουμε εντό εισαγωγικών κάπως καλύτερα σε αντίθεση με ορισμένε άλλες πρωτοβουλίες που συζητήσαμε πριν έχουμε και άλλες δυνατότητες να εφαρμόσουμε τους στόχους αυτούς και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αν δεν τους εφαρμόσουμε ε, πώς, θα, πώς θα ζητήσουμε από τους άλλους να τους εφαρμόζουν δεν είναι τόσο αξιόπιστη η στάση αυτή εάν δεν κάνουμε τα ίδια εντός με αυτά που ζητούμε να γίνουν εκτός να μπορούμε να δείξουμε δηλαδή στα Ηνωμένα Έθνη πιστικά επιχειρήματα σχετικά με το τι κάνουμε ήδη εμείς εδώ. Και κάτι από όλα αυτά, ένα από όλα αυτά βέβαια, είναι το κλίμα. Έχουμε παίξει πρωτοπόρο ρόλο και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, για την δράση για το κλίμα. Εγώ είχα καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης και αυτό ξεκίνησε όλη την ιστορία για τη Συμφωνία του Παρισιού που ήταν πραγματικά μια σημαντική στιγμή στην πορεία αυτή αλλά πρέπει τώρα να φροντίσουμε ώστε να εφαρμοστεί η Συμφωνία του Παρισιού και γνωρίζουμε ήδη ότι η Συμφωνία του Παρισιού και το περιεχόμενό της δεν αρκούν τέλος πάντων ας κάνουμε το πρώτο βήμα πρώτα και το πρώτο αυτό βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού έχουμε και νέα θέση τώρα των ΗΠΑ. Και αφού υπάρχει αυτή η νέα θέση, αυτό σημαίνει και μεγάλη ευθύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνοι μα βέβαια, αλλά σε συνεργασία με άλλου. Εδώ συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την Κίνα. Αντιθέτω από άλλου τομεί. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε πιο πολλού συμμάχου και φίλου στην προσπάθεια αυτή. Και η διπλωματία του κλίματο είναι ένα από τα εργαλεία αυτά. Προετών ήμουν Γενικό Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαμε αρχίσει ήδη να το σκεπτόμαστε αυτό το πράγμα και χαίρομαι που έχει προχωρήσει και τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Σημαντικό είναι και ο ρόλος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού το πακέτο μέτρων πέρασε πρώτα από εδώ και ενισχύθηκε από τη στάση του Ευρωκοινοβουλίου. Βρίσκω ότι υπάρχει πολύ σημαντικός ρόλος των ευρωβουλευτών και στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη. Διότι οι ευρωβουλευτές μπορούν να πούν πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι μπορεί να τα, μπορώ να τα πω εγώ ως διπλωμάτης. Και γνωρίζω ότι αυτά σκέπτεται και η κυρία Μογκερίνη και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και νομίζω ότι μπορείτε να μας ζητήσετε να συνεργαστούμε σε αυτό το συλλογικό στόχο. Δηλαδή να φέρουμε να βάλουμε σε αυτή τη συνένεση των Παρισίων περισσότερες χώρες και να προχωρήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ και Τάνοκ για την διαρκή αυτή πορτογαλοφιλία σας. Λουσιτανοφιλία λέει ο α, πρέσβης. Ε, γνωρίζω ότι είσαι από παλιά μέγας φίλος της Πορτογαλίας και μιλάτε θαυμάσια πορτογαλικά. Τώρα, Βρετανική αποχώρηση και Συμβούλιο Ασφαλεία. Για να απαντήσω και σε ορισμένε άλλε ερωτήσει για το Συμβούλιο Ασφαλεία ταυτόχρονα, μία από τι προτεραιότητέ μου αυτέ τι ημέρε είναι να ενισχύσουμε και να εντατικοποιήσουμε την συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών μας που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλεία και μεταξύ αυτών και τη δική μου ομάδα και όλων των υπολείπων που δεν είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό προβλέπεται και στη συνθήκη. Δηλαδή ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συνεργάζονται με τα μη μέλη. Αυτό που προσπαθούμε όμως να επιτύχουμε είναι ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που είναι, οι χώρες που είναι μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα εργαστούν ως ομάδα, δηλαδή τα μέλη της Ένωσης που είναι μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για να προωθήσουν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η ερώτησή σας αναφέρεται στο γεγονός ότι Εάν όλα πάνε καλά, ένα από τα δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποχωρήσει. Και τι γίνεται με τους 27 αφού θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρώπη. Θα σας πω τη δική μου οπτική χωρίς καμία απολύτω ανάμειξη στι διαπραγματεύσει για το Brexit, όπου ευτυχώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Ευτυχώ λέω. Βλέποντα τα πράγματα από την Νέα Υόρκη, είναι λογικό χώρες οι οποίες στην ουσία έχουν τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρχές. Και εγώ νομίζω και τα ίδια γεωστρατηγικά ενδιαφέροντα. Είναι λογικό λοιπόν οι χώρες αυτές στο μέλλον να βρουν τρόπους να συνεργαστούν πάρα πολύ στενά. Αυτό το έχουν πει και διάφοροι άνθρωποι και ασφαλώς θα είναι και το αντικείμενο πολύ σημαντικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Δεν θα κινηθώ περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή, απλώς λέω παρατηρώντας τα Ηνωμένα Έθνη όπως το κάνω εγώ, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο μέλλον η συνεργασία αυτή. και ούτε νομίζω ότι μπορούμε ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη να έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε διαιρεμένοι στο, στο σημερινό κόσμο. Τώρα, το πώς θα γίνει, οι τρόποι, ε, ο χρονισμός, αυτό δεν είναι δική μου υπόθεση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σήμερα και μέχρι σήμερα δεν έχω δει καμία διαφορά στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις προσπάθειες συντονισμού που κάνουμε, στις συναντήσεις μας, τα πράγματα είναι όπως πάντα. Business as usual. Και έτσι νομίζω ότι και πρέπει να είναι, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρες μέλος ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το μέλλον θεωρώ ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ στενή συνεργασία. Αλλά δεν θα πω εγώ πώς θα γίνει αυτό. Για το Κυπριακό. Στις πιο πρόσφατες συζητήσεις μας με τον Γενικό Γραμματέα ήταν σαφές ότι και ο ίδιος είναι έτοιμος και τα δύο μέρη είναι έτοιμα. Και ο ίδιο και βεβαίως και όλοι εμείς που τον υποστηρίζουμε, θέλουμε να υπάρξει λύση και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αντίθετα με την προηγούμενη φορά θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να βρεθεί λύση. Εξαρτάται βέβαια αυτό από την διαθεσιμότητα των μερών. Πιο γενικά τώρα για τις μεταρρυθμίσεις στα ΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και απαντώ εδώ και στην κυρία Γκόμες και σε άλλους. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε ο Αντώνιο Γκουτιαρές και τις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως δεν περιλαμβάνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει υποβάλει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτά συζητούνται σε ξεχωριστό πλαίσιο των χωρών μελών. Σε ό,τι αφορά εμάς, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν προβλέπουν όλες οι χώρες μέλη μας τις ίδιες λύσεις. Και όταν έχω χώρες μέλη με διαφορετικές γνώμες, είμαι αναγκασμένος και εγώ να περιορίσω το εύρος της δικής μου γνώμης και τη δική μου δράσης. Άρα, ξεφεύγει από τις αρμοδιότητές μου. Και είναι αλλιώ τα πράγματα όταν έχετε χώρε μέλη με πολύ θεμελιώδει διαφορέ μεταξύ του ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Για, για του περιορισμού του δικαίωματο ανησυχία, για δύσκολε περιπτώσει όπω η γενοκτονία για παράδειγμα, εκεί νομίζω όλοι συνυπογράφουμε. Όμω δεν συμφωνούν όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία για περιορισμού στο ΒΕΤΟ για τις προτεραιότητες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγιναν και εκεί ορισμένες ερωτήσεις οι δύο καλοί μου φίλοι εδώ στο κέντρο της αίθουσας εγώ συμφωνώ με πρόσωπα που λένε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην προώθηση που κάνουμε των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ο τρόπος με τον οποίο προσκαλούμε και άλλους να εμπλακούν σε ένα ζήτημα το οποίο είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα υπήρξαμε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Καμιά φορά κάποιες χρονιές τα καταφέρουμε καλύτερα. Αν δω την Τρίτη Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Νέα Υόρκη ή το Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Κάτι που προωθούμε μαζί με τον Σταύρο Λαμπρινίδη που είναι ειδικό εκπρόσωπο ανθρώπινων δικαιωμάτων τη κύρια Μογκερίνη είναι να φέρουμε και άλλες χώρες, ιδίως από τον Νότο, να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας αυτή, τονίζοντας τα καλά εκείνα πράγματα που κάνουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ίδιες τις χώρες τους. Άρα δεν μιλούμε μόνο για Ευρωπαίους και Καναδούς οι οποίοι, α, κοιτάξτε, λένε στον υπόλοιπο κόσμο τι πρέπει να κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να πάρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών όπου χώρες του Νότου, του Νότιου ημισφαιρίου δηλαδή, αναπτυσσόμενες, χώρες που έχουν προβλήματα ανάπτυξης, αλλά παρόλα αυτά προτάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αφήγημα ορισμένων που λένε «Α, πρώτα χρειάζεται ανάπτυξη και μετά βλέπουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Και αυτό κερδίζει έδαφος μέσα σε ένα είδος ιδεολογικής διαμάχης στην διεθνή σκηνή, όπου οι θέσεις αυτές δέχονται κάποια υποστήριξη. Μια από τις ιδέες λοιπόν που προωθούμε και πρέπει να φανούμε και δημιουργική και αναμένουμε και δική σας υποστήριξη καθώς και της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αλλά και της ΑΦΕΤ γενικότερα. Πάμε να κάνουμε κάποια πράγματα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στο μέτωπο αυτό. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, συνολικά βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Νομίζουμε ότι η Συμφωνία του Μίνσκ είναι η μόνη λύση προς, οδηγεί προς τα εμπρός. Έχει ακουστεί και η ιδέα για μια peacekeeping mission στην Ουκρανία. Ειλικρινά νομίζω ότι η διαφορά είναι τώρα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σχετικά με το πεδίο εφαρμογής ας πούμε της ε, αποστολής αυτής και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο παρόλο που το παρακολουθώ προσεκτικά για το μεταναστευτικό και βεβαίως και με ουσιώδεις διαφορές αντιλήψεων στο μεταναστευτικό που άκουσα τα τελευταία λεπτά και κάνουν πιο δύσκολη τη δουλειά μου όταν εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ζητούσα ενότητα προηγουμένω. Επ' αυτού αντιλαμβάνομαι βέβαια πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί ενότητα στο θέμα αυτό. Εμείς υποστηρίζουμε μια ε, μια πολιτική στο μεταναστευτικό επικεντρωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες των όσων είπε η κυρία Μπόξκορ. Δεν μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις εδώ και τώρα. Σε αυτό το θέμα, ο μοναδικός σκοπός που έχω, διότι στο κάτω της γραφής η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο διότι αντελήφθη ότι ε, το μεταναστευτικό δεν είναι μονάχα ευρωπαϊκό θέμα, είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα και χρειάζεται ένα παγκόσμιο πλαίσιο, παγκόσμιων λύσεων. Είχαμε την δήλωση, πολύ καλά, ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις για ένα Global Compact και για πρόσφυγες και για μετανάστες ο ρόλος μας τώρα είναι να κάνουμε την προσπάθεια αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο να απηχεί τις δικές μας απόψεις. Και γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή. Έχετε υπόψη σας λοιπόν αυτό, διότι διαιρεμένοι δεν μετρούμε στη συζήτηση αυτή. Δεν έχουμε κάποια βαρύτητα. Σε ό,τι αφορά την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Υόρκη και ο Γιώ Λάινεν ανέφερε μερικά νούμερα αρκετά εντυπωσιακά. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε ισχυρότεροι από ποτέ μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών λόγω των διαφόρων λόγων και το πώς συνεργαζόμαστε και ότι έχουμε ε, καταλάβει ορισμένε πολύ σημαντικές θέσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε περισσότερο είναι να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά μέσα στο ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας και να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε όπου αυτό είναι δυνατό, ενωμένοι γύρω από μια κοινή θέση. Αναφέρθηκα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν θέλω να αφήσω καμιά ερώτηση αναπάντητη ή σχόλιο. Κατανοώ την άποψη εκείνων που δεν θέλουν ενία έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατανοώ και τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν και τα σημειώνω. Για την ώρα σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας ξαναλέω υπάρχουν διαφορετικές θέσεις των ε, χωρών μελών αλλά γίνεται συζήτηση και εδώ και στη Νέα Υόρκη σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας σήμερα την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των χωρών. Πολλά μπορεί να πει κανείς γι' αυτά. Και τέλος για τα φορολογικά. Δεν μπορώ να πω ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεσμεύονται απολύτω υπέρ του στόχου αυτού. Υπάρχουν ίσω άλλα όργανα, αλλά δεν γίνονται πολλά πράγματα στο μέτωπο αυτό μέσα στα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Γίνονται βέβαια συζητήσει στον ΟΟΣΑ και σε άλλα φόρουμ, αλλά όχι αναγκαστικά στα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι σας κάλυψα τους περισσότερους και τις περισσότερες. Πολύ ευχαρίστως και διμερός, αν θέλετε. Ξέρετε που θα με βρείτε, όπως λένε, και όποτε θέλετε, ελάτε στη Νέα Υόρκη, αλλά ειδοποιήστε με λίγε εβδομάδε πριν, ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για λογαριασμό σα Και ξαναλέω, οι ευρωβουλευτές έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στις εξωτερικές σχέσεις και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τη συνθήκη, αλλά νομίζω και ω πολιτικοί μπορείτε να βοηθήσετε σημαντικά στην προώθηση των στόχων μας και στη διατήρηση των αξιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Ε, θαυμάσια παρουσία όπως πάντα. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται τα μέλη τη Επιτροπή μα για το τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο. Μην ανησυχείτε, θα μα έχετε. Και βεβαίω θα περάσουμε δύο-τρει ενδιαφέρουσε μέρε ε, παρέα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη ζήτηση για αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Γεια σου, Ρικάρδο. Λοιπόν, το επόμενο θέμα στην μέση διάταξη όπου θα συμπροεδρεύσουμε την Κλέα Μούντι. Είναι εδώ. Λοιπόν, ο, ο επισκέπτης μας, ο πρέσβης Ματέους Πάουλα, είναι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα στην μέσα διάταξη. Ξέρω ότι κάποιοι πρέπει να φύγετε νωρίς, οπότε θα πρότεινα να ε, μην ε, κρατήσει το επόμενο θέμα πάνω από μια ώρα, να τελειώσουμε κατά τις 11 και 4. Είναι πορτογαλική, πορτογαλικό πρωινό σήμερα στην ΑΦΕΤ. Μετά τον πρέσβη κύριο Ντεαμέιντα έχουμε τον πρέσβη κύριο Ματέου Σπάουλα, που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Δημοκρατία του Νίγηρα. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Ορισμένοι σας είδαμε ήδη στην πρόσφατη επίσκεψη στο Νίγηρα, στο Νιαμέ και το Αγκαντές. Ξέρουμε πολύ καλά την κατάσταση. Ο Νίγηρας ε, ε, είναι μια χώρα ε, πρότυπο θα έλεγα. Έχει ένα λειτουργό, λειτουργικό, δημοκρατικό, πολιτικό σύστημα. Οι πολιτικοί γνωρίζουν τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν και τι αντιμετωπίζουν. Ο Νίγηρας είναι μία από τις αφρικανικές χώρες που συνεργάζεται πολύ καλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την αποστολή μας κάψα χέλ επιτόπου και με τις γαλλικές δυνάμεις της ε, επιχείρησης Μπαρκάν. Ευχαριστώ τον πρέσβη Ματέους Πάουλα για τη στήριξη και τη φιλοξενία του κατά την κοινή αντιπροσωπή Άφετ Σέντε στο Νίγηρα πρόσφατα από την οποία εποφεληθήκαμε ιδιαίτερα. Να δώσω τον λόγο λοιπόν τώρα απευθείας στον πρέσβη. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι κάποιος από την ΣΕΝΤΕ. Όχι. Ωραία. Να δώσω απευθεία το λόγο στον πρέσβη για να ξεκινήσουμε αυτήν την αλλαγή απόψε. Για άλλη μια φορά, καλώς ήρθατε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι πολύ ευχάριστο για μένα να συμμετέχω στις ε, συνεδριάσεις σας και επίσης ήταν πολύ ευχάριστη η επίσκεψη μας κάνετε και μία άλλη αποστολή σας ε, τον Απρίλιο. Αλλά η δική μας, ε, λέει ο πρόεδρος αντιπροσωπεία, είναι πάντα καλύτερη, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, πρόεδρε. Λοιπόν, ε, λίγα λόγια για την κατάσταση επιτόπου στη δημοκρατία του Νίγηρα, Νιζέρ, που θα το συνδυάσω με τα θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης, που είναι οι δύο κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως ξέρετε, ο Νίγηρας είναι η φτωχότερη χώρα στον κόσμο. Η τελευταία στον κατάλογο με βάση τους ε, δείκτες ανάπτυξης ε, των Ηνωμένων Εθνών. Και αντιμετωπίζει και ένα τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας. Γιατί είναι ανάμεσα στο Μαλή, τη Λιβύη και ε, στο Νότο έχουμε τα προβλήματα με τον Μπόκο Χαράμ. Είναι λοιπόν πολύ δυσχερής η κατάσταση. Λόγω αυτών των συνθήκων ε, είναι σχεδόν θαύμα ότι εξακολουθεί να λειτουργεί η χώρα. Γιατί αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τρομοκρατών που διασχίζουν ε, τη χώρα και αυτό βεβαίως ε, επηρεάζει και την κατάσταση στην Ευρώπη, η κατάσταση στην περιοχή. Ξέρετε ότι εδώ και πολύ καιρό Έχουμε παρουσία στη χώρα αυτή για την καταπολέμηση της φτώχειας, για την ανάπτυξη κτλ. Αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω των θεμάτων ασφάλειας και καταπολέμησης τρομοκρατίας και λόγω των μεταναστευτικών πιέσεων ο Νίγηρας είναι χώρα μετάβαση στην Ευρώπη. Και όχι μόνο μετάβαση, πρέπει να καταλάβουμε, είναι και μια χώρα προέλευσης μεταναστών. Πολλοί από τη χώρα αυτή πηγαίνουν στην ακτή Ελεφαντοστού, το Τόγκο, γιατί έχουμε προβλήματα και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και ε, επειδή είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί και να αξιοποιηθεί η γη, πολλοί μετακινούνται. Και επίσης είναι και μια χώρα άφηξης. Ε, ε, είναι πολύ γενόδρη χώρα και υποδέχεται πρόσφυγες. Λόγω του Μποκοχαράμ 300.000 περίπου μετατοπίστηκαν στην περιοχή στο Μπερί υπάρχουν γύρω στους 60.000 πρόσφυγες από το Μαλί. Τώρα, η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη είναι φυσικά ότι πολλοί περνάνε μέσω του Νίγηρα. Πολλοί από την υποσαχάρια Αφρική διασχίζουν το Νιζέρ και περνάνε στο Αγκαντές και από εκεί φτάνουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά για τα θέματα αντιμετώπισης της μετανάστευσης. Το 2016 70.000 ε, μετανάστες διέσχιζαν ε, τον Νίγηρα, έφταναν στη Λιβύη και τα τρία τέταρτά τους κατέληγαν στην Λαμπεντούζα. Ενώ τώρα έχουμε μόνο γύρω στις 3.000 το μήνα. Πολλά λοιπόν έχουμε επιτύχει. Γιατί τα επιτύχαμε όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα. Ο πρώτος λόγος που μας ε, επέτρεψε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι υπήρχε πολιτική βούληση στη χώρα, όπως είπε και ο πρόεδρος. Ο Νίγηρας είναι πολύ καλός εταίρος της Ένωσης. Δηλαδή, ήδη πριν από την διάσκεψη στην ε, Βαλέτα, στα τέλη του 2015, είχαν καταστήσει απόλυτα σαφές ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ όλης αυτής της διακίνησης ε, ατόμων, ε, ναρκωτικών, όπλων και της τρομοκρατίας. Όλες αυτές ε, οι παράνομες ε, δραστηριότητες συνδέονται και τροφοδοτούν την τρομοκρατία. Έκαναν σωστή ανάλυση της κατάστασης και κατάλαβαν ότι υπήρχε μια τεράστια υπαρξιακή πρόκληση για τη χώρα τους και αποφάσισαν να την αντιμετωπίσουν με την βοήθεια της Ένωσης. Είχαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στη Βαλέτα και έξι μήνες πριν, το Μάιο, ε, υιοθέτησε ένα νόμο κατά της διακίνησης ε, ανθρώπων. Και επειδή ενέκριναν αυτό τον νόμο, τους κατηγόρησαν ότι το έκαναν επειδή τους πίεζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε, έχει απήχηση ε, αυτή η ε, κατηγορία επιτόπου, διότι ξέρετε ότι αυτά τα διαδίδουν οι διακινητές. Διαδίδουν αυτήν την ε, προσέγγιση. Αλλά εγώ μίλησα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της χώρας. Και ξέρω ότι αυτοί που αμφισβητούσαν αυτό το νόμο ήθελαν να καταργηθεί. Και γιατί το έκαναν αυτό, ακριβώς για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητε. Αλλά φυσικά αυτή είναι μια μειοψηφία. Γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι τη χώρα θέλουν να υπάρξει ανάπτυξη. Και ο Υπουργό ήταν απόλυτα σαφή. Μου είπε, Όχι, δεν πρόκειται να καταργήσουμε τον νόμο. Ο νόμο εγκρίθηκε γιατί εμεί θέλαμε να τον εγκρίνουμε. Διότι καταλάβαμε ότι ήταν προ το συμφέρον μα. Τον Μάιο εκείνη τη χρονιά υπήρξε μια δραματική κατάσταση. Γυναίκε και παιδιά βρέθηκαν ε, νεκροί στην ε, έρημο και ήταν πολίτες του Νίγηρα. Και αποφάσισαν ακριβώς να κρίνουν αυτό το νόμο και ζήτησαν τη βοήθεια της Ένωσης για να υπάρξει μια εναλλακτική λύση, να υπάρξει ανάπτυξη για τους πολίτες της χώρας. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Και όταν οι αρχές της χώρας αντιλήφθησαν ότι η εταιρική σχέση με την Ένωση ήταν αποτελεσματική και εγκρίθηκαν τα επίγοντα μέτρα και άρχισαν να ε, προχωρούν τα διάφορα προγράμματα. Βεβαίω δεν ήταν όλοι ικανοποιημένοι με το ρυθμό εφαρμογή των προγραμμάτων, ε, γιατί ήταν πήγοντα τα προβλήματα και ε, κάποια προγράμματα θέλουν χρόνο. Άρα θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, να επιταχύνουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων. Τώρα που ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα, συνεχίζονται καλά, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και εκτιμούν τα αποτελέσματα οι αρχές και θέλουν περισσότερη βοήθεια και για την ασφάλεια. Ξέρετε ότι υπάρχει η UCAP ε, Σαχέλ, η μη στρατιωτική ε, αποστολή που λειτουργεί από το 2011 εκπαιδεύοντας ε, το πολιτικό προσωπικό κατά της νομοκρατίας και μετά με μια, με, με μια νέα διευρυμένη εντολή για να εργαστούν για την παράτυπη μετανάστευση και για την διαμεθοριακή συνεργασία. Αυτή η συνεργασία ε, βοηθάει πολύ και υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα κατά της παράνομης διακίνησης. Είναι οι λεγόμενες κοινέ ομάδες διερεύνησης που απαρτίζονται από αστυνομικούς από την Γαλλία και την Ισπανία και κάνουν πολλή δουλειά στην ε, ε αντιμετώπιση και διάλυση αυτών των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης. Είναι πολύ καλή η συνεργασία. Και οι προποθέσει λοιπόν για την επιτυχία είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, να θεωρούν ότι τους ωφελούν τα προγράμματα, οι ίδιες οι αρχές και οι κάτοικοι της χώρα, κάτι που δεν ισχύει σε άλλε χώρες. Κλείνει το μικρόφωνο του μιλητή και δεν ακούμε τίποτα. Α, συγγνώμη. Α, ωραία, ξανανοίγει. Λοιπόν και δεύτερον, να υπάρχει ε, αποτελεσματική βοήθεια και επαρκής από την Ένωση. Γιατί δεν βοηθάμε μόνο εμείς, αλλά και τα κράτη-μέλη. Πρέπει να το δονήσω και αυτό. Έγιναν πολλές ε, επισκέψεις η κυρία Μέρκελ, ο πρόεδρος Λάοντε Τώρα και ο πρόεδρος Μακρό μας επισκέφθηκε. Ο πρωθυπουργό Τζεντιλόνι. Η κυρία Μογκερίνη ήταν η πρώτη. Ήταν η πρώτη της επίσκεψη μόλις ανέλαβε. Ήρθε στο Αγκαντές. Σαφές λοιπόν μήνυμα πολιτικής στήριξης. Στις 16 Μαρτίου θα γίνει μια πολύ σημαντική υπουργική συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών στον ΝΙΑΜΕ. Η συνάντηση που έγινε την προηγούμενη φορά στις Βερσαλίες. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και το Συμβούλιο και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος και θα έρθουν και οι χώρες G5 και οι χώρες προέλευση τη μετανάστευση, ακτή είναι Σενεγάλη και Γουινέα και η Λιβύη. Όλοι αυτοί θα συμμετάσχουν. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία και θα κατέληγα λέγοντας ότι φυσικά η τρομοκρατία είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Στη συνάντηση κορυφής του G5 στις ε, Βρυξέλλες, στις 23 ε, Φεβρουαρίου, δεσμεύτηκαν ότι θα δώσουν βοήθεια 15 εκατομμυρίων και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η βιωσιμότητα. Και ζητήθηκε εντολή για το κεφάλαιο 7 των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν είναι εύκολο γιατί δεν υπάρχει συνένεση από αυτό όπως ξέρετε. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά για την ανάπτυξη, την ασφάλεια, η συνεργασία ιδιαίτερα με τις χώρες προέλευσης για να αντιμετωπίσουμε τους διάφορους διαδρόμους να βοηθήσουμε και το, την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών ούτως ώστε αυτοί που φεύγουν από τη Λιβύη γιατί νομίζω ότι έχουν καταλάβει τώρα καλύτερα οι χώρες προέλευσης μετά από αυτά τα άθλια ε, βίντεο που είδαμε τα φρικόδη βίντεο που είδαμε στο CNN ε, άρχισαν να καταλαβαίνουν τα προβλήματα χώρε προέλευση γιατί αρνούν να τα δουν μέχρι τώρα. Τώρα υπάρχει πολύ καλύτερη συνεργασία και υπάρχει μία βούληση για να εργαστούμε, αλλά σε τελευταία ανάλυση πρέπει να έχουμε πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη ανάπτυξη, τη εκπαίδευση και το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά και με χαρά να απαντήσω ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος Μακάλιστερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Πράγματι από τις πιο ενδιαφέρουσες επισκέψεις και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε ότι ο Νίγηρας είναι από τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους εταίρους παρόλο που η χώρα αυτή είναι τόσο φτωχή. Κάθε προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τη χώρα αυτή είναι πράγματι ε, εξαιρετικά σόφρον επιλογή. Ας έρθουμε τώρα στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Έχω τέσσερα ονόματα. Πρώτος ο κύριος Πανζέρη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο σύντομες ε, παρατηρήσεις. Ήθελα τη γνώμη σας ε, και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξής. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ο Νίγηρας είναι ένα κράτος... Ε, Μ' ακούτε? Με ακούτε? Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ο Νίγηρας στην ουσία έχει σχεδόν ε, γίνει ένα νέο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η απουσία μιας κοινή πολιτικής για τη μετανάστευση έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάσταση να εξωτερικεύει τη, τα σύνορά της και άρα να εντοπίσει τον Νίγηρα ως ένα κεντρικό στοιχείο αυτής της ε, ε, εξωτερικεύσης όμως αυτό ε, συνοδεύεται από μια σειρά προβλημάτων και θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι σε αυτόν τον χώρο όσον αφορά τη μετανάστευση. Δεν υπάρχει εμφιβολία ότι στο Αγκαντές, το οποίο ήταν ανέκαθεν το σταυροδρόμι της μετανάστευσης, λειτουργήσε στο να περιορίσει την άφηξη μεταναστών, αν και ε, εξακολουθούν να έρχονται. Ορισμένοι έχουν ε, κάπως ε, μοιραστεί στην περιοχή, στην έρημο και άλλοι έχουν στην ουσία κρυφθεί, δεν τους βλέπουμε αλλά μπορεί να έρθουν σε επαφή με τους εμπόρους ναρκωτικών και όπλων που αποτελούνται κυρίως από ομάδες τζιχαντιστών που δρούν στην περιοχή. Το δεύτερο στοιχείο είναι η στρατιωτική, μεγάλη στρατιωτική παρουσία στη χώρα που κατά κάποιο τρόπο εντοπίζεται ως παρουσία για να περιορίζει το, τη μετανάστευση, και, αλλά στην πραγματικότητα ε, οδηγεί σε αντιδράσεις, γιατί αυτή η στρατιωτική παρουσία μπαίνει στο στόχαστρο των ε, αναδυόμενων ε, ε, τζιχαντιστών ηγετών όπως ο Σαράουι ως δηλαδή δυνάμεις εισβολής στη χώρα οπότε δεν τους, δεν τους θέλουν στη χώρα. Θέλω λοιπόν να έχω τη γνώμη σας αυτή η επιχείρηση που έγινε μεγαλύτερου ελέγχου της επικράτειας για να αποφευχθεί η ροή των μεταναστών αν φέρνει πραγματικά καρπούς ή αν κατά κάποιο τρόπο αποτελεί την αντικάμερα για ένα μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα ξεσπάσει στους επόμενους μήνες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα η Σιάρο Τσάλ προεδρος ευχαριστω και τωρα Ισιάρο τσαλ στανοκ Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Πανζέρη ότι τα αποτελέσματα των Ιταλικών εκλογών θα έλεγαν ότι οι ενεξέλεγκτοι ροές προσφύγων από την Υποσαχάρη Αφρική και το Σαχέλ θα είναι τεράστια, δείχνουν ότι θα είναι τεράστιες προκλήσεις για αυτές τις περιοχές και όχι μόνο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον βλέπουμε την άνοδο στην εξουσία των λαϊκιστικών κομμάτων που σαφώς ε, ε, επηρεάζουν αυτή την υπόθεση και σαφώς το τι συμβαίνει στο Σαχέλ, η σταθεροποίηση του Σαχέλ, κλιματικές αλλαγές στο μέλλον θα εξεκολουθήσουν να καταστούν την αυτό το θέμα τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις επόμενες δεκαετίες. Αλλά θέλω να εστιάσω σε μια πιο άμεση απειλή, τη, η δολοφονία ενός Αμερικανού ε, ε, στρατιώτη στον Ήγηρα τον περασμένο Οκτώβρη ήταν κάτι το οποίο έπρεπε στην αντίληψή μου και έκανα μια έκθεση στο Σαχέλ, για το Σαχέλ γενικά ως περιοχή. Ξαφνικά δηλαδή έπρεπε να εστιάσουμε σε αυτόν τον ε, αυτοκινητόδρομο θα έλεγα από τα δυτικά στα τολικά της Αφρικής για τον Μπόκο Χαράμ, ε, το Αλσαμπάμπ, και πάλι δηλαδή πρόκειται για έναν ε, δρόμο μέσω του οποίου ε, οργανώνονται όλα τα εμπόρια, τα παράνομα εμπόρια ναρκωτικών, όπλων, ανθρώπων και αποσταθεροποιείται έτσι όχι μόνο η Αφρική αλλά έχει και παγκόσμιο αντίκτυπο το τι γίνεται εκεί. Η δε συνεχιζόμενη ήττα ε, του ISIS στη Συρία και στο Ιράκ ε, σημαίνει πως ε, θα, προχω... θα έρθουν προς αυτή την περιοχή και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν ε, οι τζιχαντιστές. Ο καθορισμός των συνόρων δε σε ορισμένες χώρες του Σαχέλ είναι πολύ δύσκολος γιατί στην ουσία είναι σύνορα χαραγμένα στην άμμο. Γίνονται περισσότερα ώστε να οριοθετηθούν οι χώρες και να ελεγχθεί καλύτερα η κίνηση των ανθρώπων, ειδικά των τρομοκρατών και του, οργανωμα... οργανωμένου Και κάτι ακόμα θυμάμαι από την έκθεση για τον Νίγηρα. Ο Νίγηρας έχει μεγάλα κοιτάσματα ουρανίου που βεβαίως ε, θα ήταν ε, καταστροφικός στόχος για τους διεθνείς τρομοκράτες αυτός, εάν δηλαδή έβαζαν τα χέρια τους αυτά τα κοιτάσματα και άρχισαν να εξάγουν σημαντικές ποσότητες. Είναι ένα διενεργό, αν όχι πυρηνικό όπλο, αν φτάσει στην Ευρώπη. Είναι ασφαλισμένα τα ορυχεία ουρανίου στον Ήγηρα ε, εναντίον τέτοιων προσπαθειών. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέζινγκ της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα, εντάξει έχετε τα ακουστικά σας, ωραία. Πρόσφατα λοιπόν λέγω, εδώ βρίσκομαι κύριε Πρέσβη εκεί πίσω. Πρόσφατα λέω είχαμε μια high level conference Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής όπου μπορέσαμε να ακούσουμε πολλές πληροφορίες και από τον Νίγηρα. Η κατάσταση εκεί είναι πολυεπίπεδα προβληματική και όταν βλέπουμε την κατάσταση και μέσα από τα μάτια των χωρών αυτών γι' αυτό μας βοηθεί να αποφύγουμε να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα επιπρόσθετα των υπαρχόντων. Ένας άνθρωπος λοιπόν από τον Ήγηρα μας εξήγησε τα πράγματα αυτά με πολύ ανάγλυφο τρόπο ότι δηλαδή το διαμεθοριακό εμπόριο στη χώρα αυτή είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο παραδοσιακό και πάρα πολύ διαδεδομένο και από, τα πιο, ε, από τις πιο σημαντικές πηγές βιοπορισμού για τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για παράνομο εμπόριο και τρομοκρατία και ε, σωματεμπορία κτλ. Αλλά είναι όλο αυτό μέσα, μπλεγμένο μέσα σε ένα πάρα πολύ περίπλοκο και πολυσχηδές επιχειρηματικό μοντέλο. Ε, η ερώτησή μου είναι για το Σαχέλ. Ε, λαμβάνεται υπόψη αυτή η ευρεία βάση βιοπορισμού και τι επιτυχία αναμένεται από κάποιες προσφορές αντιστάθμισης και αν μπορείτε να κάνετε κάποια αποτίμηση αυτών των δυνατοτήτων αντιστάθμισης. Εμάς μας είπαν Μα είπαν ότι εκεί πρόκειται για κάτι σαν ατμολέβητα που ετοιμάζεται να εκραγεί η χώρα αυτή δηλαδή, το, ο Νίγηρας. Και από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών μας είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και ο ίδιος ο Νίγηρας λέει ότι δεν θα δεχτεί άλλους πρόσφυγες εάν δεν μπορεί να τους παροχετεύσει περαιτέρω ε, προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγαλύτερο βαθμό. Μιλήσατε και για τους θανάτους στην έρημο. Στο κρατικό κανάλι ARD στη Γερμανία, σε μια εκπομπή είδα ότι στρατιώτες του Νίγερα έχουν τοποθετηθεί μετά από προτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σημεία ανεφοδιασμού με νερό των προσφύγων που περνούν από την έρημο για να τους εμποδίσουν να πάρουν νερό από τις πηγές αυτές και τελικά οι άνθρωποι πεθαίνουν από τη δίψα. Και μια ερώτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διεθνής Αμνηστία μας είπε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους πρόσφυγες είναι εξαιρετικά δεινή. Πώς είναι λοιπόν δυνατό υπό τις συνθήκες αυτές να παρατηρηθούν οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στη χώρα αυτή στην Ήγυρα. Πώς εκτιμάτε εσείς την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, τρομοκρατία και αποσταθεροποιητική ενέργεια το G5 και μιλήσατε και για την ανάγκη αηφορίας της παρέμβασης αυτής. Τώρα, μάλιστα την προηγούμενη Παρασκευή, σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο σε μια επίθεση 20 άνθρωποι που είπαν ότι ήταν αντίδραση η επίθεση αυτή της Αλκάιντα στην αποστολή του G5. Ανησυχώ πολύ λοιπόν. Κατά πόσο δηλαδή με την παρέμβαση του G5 ε, έχει ξεκινήσει ή μπορεί να ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος ο οποίος θα οδηγήσει όλο και περισσότερο σε μια αποσταθεροποίηση Και τέλος, ερώτηση κατά την άποψή σας πόσο υψηλό είναι το κόστος, το τρέχον κόστος της αποστολής των G5 στην Σαέλ. Κάτι άκουσα για 150 εκατομμύρια και διαρωτώ με από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Λέζινγκ. Ο κύριος Μπούχνερ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι στο τελευταίο που είπατε. Είπατε ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνίσταται ιδίως σε αναπτυξιακή βοήθεια, εκπαίδευση, παιδεία δηλαδή, και απασχόληση και το δημογραφικό. Περισσότερες λεπτομέρειες, ιδίως για την αναπτυξιακή βοήθεια, όπου σε πολλές αφρικανικές χώρες η αναπτυξιακή βοήθεια ναι μεν βοηθεί σε ένα πρώτο πλάνο αλλά ταυτόχρονα συνδέεται με περιορισμό κάποιων δικαιωμάτων καλλιέργειας. Με ενδιαφέρει λοιπόν ποια είναι η επίπτωση της αναπτυξιακής βοήθειας ιδίως στον αγροτικό τομέα. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Δεν έχω άλλα σχόλια. Προσπαθήστε κύριε Πρέζη να απαντήσετε. Μία παρατήρηση δική μου, διότι η κυρία Λέσινγκ επεκτάθηκε ιδιαίτερα για τις παρεμβάσεις των δυνάμεων της G5. Πήγαμε επί τόπου και η δική μου πάντως εντύπωση ήταν ότι από όλου τους συνομιλητές μας ακούσαμε επένους και έκφραση ευγνωμοσύνης για την δέσμευση αυτή, γιατί είναι εμπλοκή μα αυτή και ότι ο αγώνα κατά των τρομοκρατών είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή και ότι οι τρομοκράτε έχουν καταστρέψει τις Αγκαντέ τη βάση διαβίωση των ανθρώπων ενώ οι Αγκαντέ παλιά ήταν η πόρτα προ την έρημο και για Ευρωπαίου και Αμερικανού που ήθελαν να επισκεφθούν την έρημο όλο αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο που βασιζόταν στου περιηγητές αυτού κατέρευσε. Εγώ πάντως επενώ μεγάλο την γαλλική στρατιωτική παρέμβαση επιτόπου που ηγούνται αυτής της, ε, που ηγείται μάλλον αυτή τη προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας που είναι εξαιρετικά εύστοχες. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω κάπως τη σειρά με τις οποίες ετέθησαν οι ερωτήσεις. Καταρχάς, η εξωτερήκευση των συνόρων. ότι δηλαδή η Ένωση έχει τοποθετήσει τα σύνορά της στον Νίγηρο εφόσον στην Λιβύη η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεν υπάρχει κυβέρνηση, μάλλον υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις, πολύ περίπλοκη κατάσταση. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει πάντως να δώσουμε περισσότερες αποχρώσεις. Είναι προφανές ότι ο Νίγηρας έχει καταστεί εξαιρετικά σημαντικός εταίρος για την Ένωση, διότι είναι σαφές ότι η γεωστρατηγική θέση της χώρας παίζει ρόλο προφανώς λόγω των θεμάτων ασφαλείας ε, που αναφέρθηκαν ήδη, τρομοκρατία, νομίζω πως η τρομοκρατία, την τρομοκρατία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για το Σαχέλ, για τον Νίγηρα, για την Ευρώπη. Διότι είναι ε, στη πρόθυρα. Είναι είναι στην ουσία τα σύνορα της Ευρώπης ε, ε, και πρέπει αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, εδώ στον Ήγηρα έχουμε την ε, τύχη, το θυμίζω και νομίζω το υπογράμμισε και ο πρόεδρος. Έχουμε την τύχη να έχουμε έναν εταίρο αξιόπιστο. Έναν εταίρο που ακόμα και αν είναι η πιο φτωχή χώρα του κόσμου, είναι ε, ε, ιδιαίτερα περήφανοι για την κυριαρχία τους και αυτό το έχουν επιβεβαιώσει πολλές φορές. Δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τα ασφάλματα που έχουν γίνει αλλού. Για παράδειγμα, είδατε τι έγινε λίγο στο Μαλί. Τότε ο πρόεδρος σιγά σιγά υποχώρησε και η κυβέρνηση δεν ήταν ε, παρούσα. Ε, είδατε ποιο ήταν ε, το αντίκτυπο για τη διεθνή κοινότητα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακτήσουμε την κυριαρχία του κράτους αυτού. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Στον Ήγερα είμαστε σε διαφορετικό πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μεγάλη συνύπαρξη. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργό είναι του Αρέγκα Μόλις όρισε τον επικεφαλής του επιτελείου του στρατού, του Αρέγ επίσης. Υπάρχει δηλαδή μια συνοχή, μια πολύ έντονη θέληση. Τώρα, για το θέμα της στρατιωτικής παρουσίας. Οι Γάλλοι είναι παρόντες με την επιχείρηση Μπακράν εδώ και καιρό. Ε, είναι προφανές ότι ζήτησαν από τους Ευρωπαίους εταίρους αλληλεγγύη και νομίζω πως αυτή η φωνή εισακούστηκε. Πρέπει να πω για παράδειγμα η Γερμανία είναι όλα και πιο παρούσα στον Ήγηρα και στο Σαχέλ. Υπάρχει στρατιωτική συνεργασία, ενώ προηγούμενα υπήρχαν οι Γάλλοι μόνο και οι Αμερικανοί, που είναι επίσης πολύ παρόντες, ιδιαίτερα παρόντες στον Ήγηρα και στην ανάπτυξη και στην, ε, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και η Ιταλία έφτασε. Έχουν γίνει επιχειρήσεις, ε, τώρα γίνεται εξολόγηση με Ιταλούς στρατιωτικούς ώστε να γίνει η κατάρτιση. Και βεβαίως ε, υπάρχει και η πολιτική συμφων... αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΟΚΑΠ. Βεβαίω, υπάρχουν αντιδράσεις ε, του πληθυσμού, αυτό είναι προφανές, είναι πολύ λεπτό θέμα η παρουσία στρατιωτικών βάσεων. Η παρουσία αυτή απαιτεί προσπάθειες από πλευράς της κυβέρνησης και του Προέδρου Ισουφού, δηλαδή προσπάθειες εξήγησης το τι συμβαίνει. Κάθε φορά θυμίζει λοιπόν, το κάνει αυτό ο Πρόεδρος και κάθε φορά θυμίζει την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία των συμμάχων, γιατί η τρομοκρατία είναι πραγματική απειλή. Το είδαμε στην Μπουργκίνα Φάσο πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα. Η τρομοκρατία χτυπά παντού, στο νεκριτή του ελεφαντιστού, στο Μαλί επανελειμμένα. Στον Νίγηρα λοιπόν το πρόβλημα έρχεται από το Μαλί και από τη Λιβύη και βεβαίως και από το Μπόκο Χαράμ που δεν είναι υπό έλεγχο ακόμα. Τρία είναι τα μέτωπα δηλαδή στα σύνορα, αλλά το κράτος στον Νίγηρα λειτουργεί. Είναι ένα κράτος και γι' αυτό και μαζί τα βοήθεια και τα λοιπά. Έχουν ε, και καλές μυστικές υπηρεσίες και καταφέρνουν να προλάβουν πολλές απόπειρε. Όμως ο Νίγηρας αυτή τη στιγμή είναι ο προεδρεύει του G5 Σαχέλ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλά τη σχέση ανάμεσα στην ε, ασφάλεια και την ανάπτυξη δυνάμεων. Στο Μάντι, στο κέντρο λοιπόν, ανάμεσα στο Μαλί, τον Νίγηρα και την Πουρκίνα Φάσο, έχουμε εξαιρετικά αποσταθεροποιημένη ζώνη και όλα τα προβλήματα έρχονται από το μαλλί, από την αποσταθεροποίηση του μαλλί εκεί. Για παράδειγμα, έχουν δολοφονηθεί εκεί καθηγητές. Δηλαδή θα βρείτε παιδιά που δεν μπορούν να πάρουν σχολείο. Γιατί οι καθηγητές φοβούνται. Καταστάσεις που πραγματικά εφόσον δεν υπάρχει ασφάλεια δεν, ασφάλεια, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Οι απειλές είναι πολύ πολύ έντονες. Υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση που επίσης στρέφεται από τη φτώχεια. Ε, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι οι απαντήσεις είναι περίπλοκες. Ναι, ασφάλεια και ανάπτυξη. Και από τα δύο χρειάζονται. Πρέπει να επιτεθούμε στις βαθιές ρίζες της φτώχειας. Να πω δύο λόγια για την ε, παιδεία στον Ήγηρα, που είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν μαζικές επενδύσεις στην παιδεία, διότι λόγω του δημογραφικού προβλήματος, του ποσοστό γονιμότητας και ανάπτυξης στον Ήγηρα είναι το πιο ψηλό στον κόσμο. Εγώ δεν θέλω να είμαι αρνητικό γιατί δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν για παράδειγμα, ο πρόεδρος Ιουσουφού και εμείς έχουμε παίξει ρόλο, οι πρέσβει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διεθνή κοινότητα έχουμε ενθαρρύνει να ψηφιστεί ένα διάταγμα για, την, ε, για τα κορίτσια και για την ε, εκπαίδευσή τους. Η δημογραφία είναι η ίδια και όλες οι μουσουλμανικές χώρες, όλες οι αραβικές χώρες έχουν καταφέρει την δημογραφική μετάβαση. Δεν είναι κάτι το αδύνατο. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν σε αυτό το τομέα. Στον Νίγηρα λοιπόν με το σημερινό ποσοστό της δημογραφίας πρέπει να κατασκευάζονται 6.000 τάξεις το χρόνο για να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο. Είναι αδύνατον. Ε, alors qu'est-ce qui s'est passé Ils ont investi, euh, ils ont investi dans l'éducation au niveau quantitatif Euh, λοιπόν, πρέπει να, ε, έπρεπε να προσληφθούν δάσκαλοι που δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Ε, πρέπει να μάθουν τα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν. Χάρη στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις αρκετά θαραλές. Ο υπουργό Παιδείας έχει, κάνει, ξεκινήσει μάλλον αξιολογήσεις για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι. Είναι τεράστια δουλειά ε, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην ασφάλεια των τροφίμων. Ε, υπήρξε και ερώτηση για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ε, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σας πω πως ο Νίγηρας είναι η χώρα που ωφελείται περισσότερο από την βοήθεια ανακάτοικο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. 600 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί με την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ε, ε προσθέθηκαν 80 εκατομμύρια ακόμα ε, και αυτά ε, χέρι με χέρι με την διατροφική βοήθεια και ασφάλιση. Με καλή διακυβέρνηση. Ε, πρέπει όλα αυτά βεβαίως να συμβαδίζουν. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, οι παρεμβάσεις μας είναι περίπλοκες και έχουμε τα επίγοντα ε, βραχυπρόθεσμα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά και τα μακροπρόθεσμα προβλήματα. Πρέπει να δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν πρέπει να χάσουμε την ε, ελπίδα μας. Είναι όμως γενικά η Αφρική είναι πολύ ζωντανή και ζωηρή ε, Ήπειρος. Ε, κινούνται τα πράγματα. Υπάρχει, υπάρχουν πολλοί νέοι, έχει γίνει ψηφιακή επανάσταση, ο κόσμος συνδέεται ε, και τους ε, σπρώχνει αυτό να θέλουν καλύτερη ζωή. Υπάρχει μεταναστευτική πίεση κλιματικές αλλαγές είναι τεράστια πρόκληση και συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Η πίεση αυτή θα συνεχίσει και πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό το τομέα. Στον Ήγηρα υπάρχει ένα πρόγραμμα για την ανάκτηση των γεών, γιατί προχωράει έρημος και πραγματικά είναι πολύ περίπλοκο, αλλά με τα κονδύλια για τις κλιματικές αλλαγές πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο σε αυτό το τομέα. Άλλη πρωτοβουλία για την Ιγυρία συγγνώμη για τον Ήγηρα, ε, είναι αυτή που, ε, αφορά το νερό για το διαμεθοριακό εμπόριο. Βεβαίως υπάρχουν, ε, υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες, λαθρεμπόρια, υπάρχουν εγκληματίες οι οποίοι κάνουν και διακίνηση ατόμων, τους παρατάνε στην έρημο, ξέρουν ότι θα πεθάνουν. Ξέρετε, αν μιλήσετε με τους μετανάστες, όπως έχω μιλήσει εγώ, έχω επισκεφτεί διάφορους καταβλισμούς Ακούτε τρομερές ιστορίες, ιδιαίτερα δραματικές, φρικώδεις. Δεν χρειαζόντουσαν τα βίντεο του CNN που πραγματικά σκανδάλισαν την κοινή γνώμη. Αν μιλήσεις με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ξέρεις πόσο οδυνηρές είναι αυτές οι καταστάσεις. Πρέπει να κάνουμε πολλά και στο επίπεδο της επικοινωνίας, πιστεύω. Γιατί αυτές οι ιστορίες που μας διηγούνται, τα δράματα που έχουν ζήσει, μπορούν να βοηθήσουν να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και μπορούν να αποτρέψουν και άλλους να ξεκινήσουν ε, παρόμοιες διαδρομές. Αλλά πρέπει να επιτεθούμε στους τρομοκράτες, στους διακινητές και πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη. Μόνο αν υπάρχει ανάπτυξη θα υπάρξει λύση. Αυτή είναι η λύση. Αλλά είναι δύσκολο. Γιατί πρέπει να δράσουμε και βράχη και μέσο και μάκρο πρόθεσμα. Αλλά είμαι πεπισμένο ότι είναι προ το συμφέρον τη Ένωση. Γιατί αλλιώ θα υπάρχουν πάντα αυτέ οι μεταναστευτικέ πιέσει. Θα συνεχιστούν θα συνεχιστούν τα προβλήματα τρομοκρατίας. Οπότε πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την ανάπτυξη. Ήδη κάνουμε πολλά. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε και προσέγγιση. Να βγάλουμε διδάγματα. Για παράδειγμα υπάρχει αυτή η κοινή δύναμη του Z5. Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι εκεί. Είναι πραγματικά αναγκαία. Γιατί υπάρχουν πραγματικές απειλές πρέπει να στηρίξουμε. Πρέπει να γίνει μόνιμη. Υπάρχουν οι τρομοκράτες που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, από τη Συρία, από το Ιράκ κτλ. Και ξέρουμε, ξέρουμε, έχουμε πληροφορίε. ότι εγκαθίστανται στη Λιβύη και στο Σαχέλ. Τρομερές προκλήσεις λοιπόν. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η βοήθειά μα Πιστεύω ότι η Ένωση είναι ιδιαίτερο παρούσα, όλο και περισσότερο και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε πολλά γιατί έχουμε υποδειγματική συνεργασία με τα κράτη-μέλη επιτόπου. Με τα καταπιστεύματα που έχουμε, η Γερμανία συμβάλλει, οι βόρειες χώρες. Και τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τα ανέφερα μέχρι τώρα. Ακριβώς. Όταν είχαμε τη συνάντηση κορυφής του G5, η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία οργάνωσαν ένα σεμινάριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινή δύναμη αυτή, τον ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εκπαίδευση της αστυνομίας για αυτά τα θέματα. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση και υπήρξε καλή βούληση συνεργασίας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι επιχείρησα... Α, ναι, α, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Για το, τα ορυχεία τώρα, τα ορυχεία ουρανίου. Ξέρετε, ο προπορισμός του Νίγηρα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ο προπολογισμό ε, ε, κατά 18% ε, αφιερώνεται στην ε, ασφάλεια. Παρά τη δική μας βοήθεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι από την άλλη μεριά κατέρευσε η τιμή του ουρανίου που συνέβαλε πολύ στον προπολογισμό. Έχουν επίσης πετρέλαιο, αλλά και εκεί κατέρευσε η τιμή. Το εμπόριο με την Ιγυρία ήταν επίσης πολύ σημαντικό, αλλά έχουμε κρίση στην Ιγυρία. Και εδώ λοιπόν κατέρευσαν τα έσοδα. Πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το ουράνιο, η Αρέβα είναι παρούσα, η γαλλική εταιρεία. Βέβαια μειώθηκαν οι επενδύσεις τους, γιατί δεν είναι επικερδές ε, πλέον, ε, δεν είναι επικερδής η εξόριξή του. Οπότε αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουμε καθόλου κρατικά έσοδα από την εξόριξη ουρανίου. Αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τις εγκαταστάσεις. Αλλά είναι, πιστεύω, Υπάρχει καλή προστασία αυτών των εγκαταστάσεων. Υπάρχουν οι γαλλικέ στρατιωτικέ δυνάμει και οι Αμερικανοί που αυτή τη στιγμή χτίζουν μια βάση στο Αγκαντέ και ενισχύουν την παρουσία του. Και για του Αμερικανού ε, στρατιώτε, ξέρετε, τέσσερι ε, δολοφονήθηκαν σε μια ενέδρα. Βεβαίω, αυτό ήταν ένα δράμα, αλλά νομίζω ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή ενισχύουν τη στρατιωτική του παρουσία. Δεν αποσύρονται, ενισχύουν την παρουσία του. Ακριβώ επειδή χτίζουν και μια βάση στο Αγκαντέ. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω, ξέχασα τίποτα. Προσπάθησα να απαντήσω σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να θέσει περαιτέρω ερωτήσεις. Όχι. Ωραία. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας και τη δουλειά που κάνετε στο Νιαμέι και νομίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα δώσουν συνέχεια στις επισκέψεις μας. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η χώρα στην οποία εκπροσωπεί την Ένωση. Επόμενο θέμα, τα διάφορα. Όχι, ωραία. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 12 Μαρτίου, Δευτέρα απόγευμα στο Στρασβούργο και να σας ενημερώσω ότι εκτός από την ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Γιάγκλαντ, θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων και για την ε, κρίση για την παροχή αερίου στην Ουκρανία. Έχουμε καλέσει εκπροσώπους από την Επιτροπή, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και επίσης τον επικεφαλής της επιχείρησης Ναύτα Γκάς Ουκρανίας. Ολοκληρώνω τη εργασία μας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.